είναι λοιπόν τα συνοπτικά πρακτικά. Ερχόμαστε στι ανακοινώσει. Οι αρμόδιε αρχέ τη ε, Ομοσπονδιακή Δημοκρατία Γερμανία με ενημέρωσαν για την εκλογή τη κυρία Γκαμπριέλη Στάουνερ από τι 30 Οκτωβρίου και τη κυρία Μπράιερ από την 31 Οκτωβρίου 2013. Ε, η κυρία Στάουνερ αντικαθιστά την κυρία Βάι Γκέρμπερ, ενώ η κυρία Μπράιερ την κυρία. Ε, Μπραντνερ, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 για τις εκλογές των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα επίσης και το άρθρο 4 παράγραφη, 1 και 4 του κανονισμού του Κοινοβουλίου σημειώνουμε την εκλογή της κυρίας Τάουνερ και της κυρίας Μπράιερ με τις αντίστοιχες ημερομηνίε γιατί λαμβάνουμε υπόψη. Καλωσορίζω τις συναδέλφους και θυμίζω ότι και η κυρία Στάουνερ και η κυρία Μπράιερ σύμφωνα ε, με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού θα συμμετέχουν ε, με πλήρη δικαιώματα ε, στα όργανα του Κοινοβουλίου μέχρι να εγκριθεί ή να προσβληθεί εντολή τους και με την προϋπόθεση ότι προηγουμένως έχουν δηλώσει ότι δεν κατέχουν κανένα αξίωμα που είναι συμβίβαστο με το αξίωμα του Ευρωβουλευτού. Οι αρμόδιες πολωνικές αργές έχουν υποβάλει αίτημα για άρση ασυλίας του κυρίου και Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού διαβιβάζεται το αίτημα αυτό ε, στην Αρμόδια Νομική Επιτροπή ε, από ε, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και την Ελευθερία και Δημοκρατία έχουν υποβληθεί